Λοιπόν, γεια σας. Ε, ξεκινήσαμε σήμερα στην ομάδα της ε, Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια μεγάλη συνάντηση, διεθνή συνάντηση ε, για την ανάγκη αλληλεγγύης ανάμεσα στις πόλεις και στις χώρες, ιδιαίτερα αυτές που δέχονται τα κύματα των προσφύγων. Στο επίκεντρο φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα και βρέθηκε και η Λέσβος καθώς επίσης και μια σειρά από άλλες πόλεις ε, που και νησιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ήταν μαζί μας η αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης που μίλησε επίσης. Ήταν ο, δήμαρχος ε, Κιλίνης και Ανδραβίδας ε, που είναι Σύριος. Ήταν η δήμαρχος της Τήλου και ήταν βεβαίως και ο κύριος Γαλινός, ο κύριος Γαλινός, ο δήμαρχος της Λέσβου, ε, ο οποίος ε, μίλησε σε αυτή την εκδήλωση. Τον έχουμε και σήμερα μαζί για να μας μιλήσει για την, ε, για την κατάσταση στο νησί, που συνεχίζει να δέχεται προσφυγικές ροές και να αντιστέκεται με μικρή βοήθεια και μεγάλες χαμένες ελπίδες και υποσχέσεις από την πλευρά της κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν όμως μας, πει, ο, μας μιλήσει ο κύριος Γαλινός, θα δώσω το λόγο στον ε, Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μας πει δύο λόγια. Ε, σας ευχαριστώ. Συνηθίζουμε να λέμε και σωστά ότι οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Υπάρχουν όμως μερικές φορές που οι αριθμοί λένε πάρα πολλά ε, για τους ανθρώπους ειδικά όταν πρόκειται για δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καταφτάνουν κυνηγημένοι με τις οικογένειές τους από εμπόλεμες ζώνες, εκεί οι αριθμοί λένε πολλά. Η Λέσβος δεν είναι απλά ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, από τα ομορφότερα ελληνικά νησιά. Είναι ένα νησί με 85.000 πληθυσμό που το 2015 δέχτηκε 500.000 πρόσφυγες. Και μέσα στο 2016 από τους 170.000 πρόσφυγες περίπου που έχουν φτάσει στην Ελλάδα, οι 95.000 έχουν περάσει ή βρίσκονται ακόμη στη Λέσβο. Η δημοσιότητα που πήρε το νησί, η μεγαλοσύνη και η ανθρωπιά των ντόπιων των κατοίκων του, η φιλοξενία των κατοίκων της Λέσβου και η ανθρωπιά τους έγιναν εξώφυλλα εφημερίδων σε όλο τον κόσμο. Πρωτοσέλιδα πολλών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωση, αλλά δυστυχώς δεν φτάνουν. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανασκουμποθεί για ολόκληρη την Ελλάδα και την Ιταλία και κυρίως για τη Λέσβο που σηκώνει στις πλάτες της δυσανάλογο βάρος. Η μετεγκατάσταση των προσφύγων προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς λόγω της έμπρακτης αδυναμίας ή και άρνησης να υλοποιηθεί μια συμφωνία που έχει ληφθεί. αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρνησης αρκετών κρατών μελών. Και η Λέσβος είναι θύμα μιας αδύναμης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών μελών που περιφρονούν τις κοινέ αποφάσεις με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παραμένουν σε αντίξωες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες στη Λέσβο και στην Ελλάδα συνολικά περίπου 60.000. Ε, η σημερινή συνέντευξη τύπου, όπω και η πρωτοβουλία που οργανώνεται από το πρωί με τα χαρακτηριστικά που σα υποστέλει ο Κούλογλου, είναι μία ακόμη προσπάθεια να ενώσουμε τι φωνέ μα για άμεση εφαρμογή τη απόφαση για μετεγκατάσταση από όλα τα κράτη-μέλη. Με το άνοιγμα από τα κράτη-μέλη των θέσεων που τους έχει οριστεί. Περίπου 10.000 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω, είναι έτοιμοι να φύγουν από την Ελλάδα και να μετεγκατασταθούν αλλά αυτό μπλοκάρεται από την άρνηση κρατών μελών. Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να μειωθεί, να εξαφανιστεί αυτή η απορριπτική απόφαση από διάφορα κράτη-μέλη που αρνούνται να δεχθούν πρόσφυγες χωρίς καμία σοβαρή δικαιολογία, να ενισχυθεί άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να έλθει και να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του ασύλου. Έχουν αποφασίσει να στείλουν 400, έχουν στείλει πάρα πολύ λίγους, ελάχιστες δεκάδες, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αλλά με σωστή εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προδιαγραφών. Και επιπλέον χρειάζεται πρόνοια και ενισχύσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα και ειδικά στη Λέσβο, να βρεθεί τρόπος να φιλοξενούνται σε καλύτερε συνθήκες τα παιδιά, τα συνόδευτα παιδιά, με έναν τρόπο που να συνάδει με συνθήκε ανθρωπιά, επομένω το σχήμα υλοποίηση των συμφωνημένων από όλα τα κράτη-μέλη, γρήγορη και ασφαλή μετεγκατάσταση, σύμφωνα και με την ποσόστοση, η ειρηνική συμβίωση με τους ντόπιου και ασφαλής μπορεί να περιορίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι πρόσφυγες αλλά και οι κάτοικοι της Λέσβου που σηκώνουν ένα υπέρογκο βάρος. Ε, η ελληνική κυβέρνηση πιέζει για ταχύτερες διαδικασίες, αξιοποιεί όσο μπορεί καλύτερα τα ευρωπαϊκά ταμεία προς αυτή την κατεύθυνση και θέλω εδώ να υπογραμμίσω κάτι, επειδή γύρω από αυτό γίνεται και μια σπέκουλα πολλές φορές. Τα περισσότερα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα λόγω των κανονισμών της Κομισιόν δίνονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Πατιαρμοστία κλπ. και όχι απευθείας στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική διοίκηση. Επομένως, εκτός από την ελληνική διοίκηση πρέπει και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να προσφέρουν περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σταματήσω εδώ και να πω ότι χαίρομαι γιατί ε, αυτή η πρωτοβουλία που οργανώθηκε ε, έχει μια μεγάλη διεθνή συμμετοχή και ε, συμπαράσταση από ευρωβουλευτές, από ένα ευρύ φάσμα χωρών, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι μόνη πριν από ένα μήνα περίπου, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με μια μεγάλη πλειοψηφία το αυτονόητο ότι θα πρέπει επιτέλους τα κράτη-μέλη να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί και να μην σηκώνουν μόνες τους το βάρος η Ελλάδα κυρίως και δευτερευόντως η Ιταλία. Ωραία, το λόγο έχει ο, ο Δήμαρχος Λέσβου. Εν αρχή θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σε μια κρίσιμη στιγμή και για τη Λέσβο και για την Ελλάδα να ενισχύσω, να δυναμώσω τη φωνή της Λέσβου μια και πριν από λίγες ημέρες έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό ε, υπό την έννοια ότι θεωρούμε ότι κάποιες κυβερνήσεις στην Ευρώπη απεδείχθησαν κατώτερες των περιστάσεων ίσως δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και τους κινδύνους που εγκυμονούνται για την ίδια την Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο ζητώ, έχω αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και ζητώ το έλλειμμα των ηγησιών να το καλύψουν οι Δήμοι, οι τοπικές κοινωνίες. Σε μια προσπάθεια και σε μια λογική ότι όταν ένα βάρος το σηκώνει ένα είναι δυσανάλογα μεγάλο και δεν τα καταφέρνει, όταν όμως το ίδιο βάρος το σηκώσουν πολλοί, τότε το βάρος εκμηδενίζεται και γίνεται ασήμαντο. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει από την Ελλάδα και έχω κάνει αυτή την πρόταση και προς την ΚΕΔΕ και προς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες δημάρχους, αλλά παράλληλα το ε, έδωσα να το επικοινωνήσω και προς την Ευρώπη. Έχουμε αρχίσει μια συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Δήμους και σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διότι έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί περισσότεροι δήμοι στην Ευρώπη και να διαπιστώσω κι εγώ ότι από πλευρά των Δήμων αυτών, πολλών Δήμων, υπάρχει διάθεση να σηκώσουν βάρος, να βοηθήσουν και εκείνοι, αλλά του εμποδίζουν οι κυβερνήσει του. Θεωρώ λοιπόν πράγματι ότι η πρόσκλησή σας ήρθε την κατάλληλη στιγμή και θα βοηθήσει πάρα πολύ να ξεμπλοκάρει αυτή η διαδικασία που μόνο κινδύνω συγκυμονεί για την Ευρώπη, που πρέπει να καταλάβει ότι ο πραγματικός κίνδυνος ή η πραγματική κίνδυνη που διακυβεύονται σήμερα από τον τρόπο διαχείρισης μιας προσφυγικής κρίσης είναι ότι αυξάνονται αλματοδός οι δυνάμεις, οι ρατσιστικές δυνάμεις και φωνές, οι οποίες όμως οδηγούν στην ενδυνάμωση φασιστικών κινημάτων. Ήδη, ε, και αυτό το έλεγα από πέρυσι και βλέπω δυστυχώς να δικαιώνομαι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση για μια αρνητική εξέλιξη, βλέποντας ότι σε εκλογικά αποτελέσματα σε διάφορες χώρες πραγματικά ακροδεξιά έως φασιστικά κινήματα δυναμώνουν και δυναμώνουν επικίνδυνα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθεί η Ευρώπη, να αντιληφθούμε όλοι μας και να δούμε ότι η πραγματική κίνδυνη δεν είναι οι άνθρωποι στους οποίους υψώνουμε τα τείχη, αλλά οι ιδέες οι οποίες στην ουσία κατασπαράζουν τις άρκες των κοινωνιών μας και τον συνδετικό του συστό. Ε, Ήδη η Ευρώπη έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τέτοιες ιδέες και τέτοιες πρακτικές. Ας βάλουμε φραγμό σήμερα, να μην το πληρώσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε Δήμαρχε. Παρακαλώ ε, υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο, στο νησί από πλευράς ε, ε, ροών που συνεχίζονται, έστω και μειωμένες, αλλά υπήρξαν κάποια, κάποιες αντιδράσεις ε, κατοίκων που φαίνεται να, ήταν υποκινούμενες. Μπορείτε να μας πείτε λίγα παραπάνω πράγματα για την κατάσταση στο νησί. Θα σας πω ότι σήμερα στο νησί υπάρχει ένα, όπως αναφέρατε και εσείς, ένα δυσανάλογο βάρος. Φιλοξενούνται περίπου 6.500 άτομα ε, σε δύο χώρους, οι οποίοι, σε τρεις χώρους, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 3.500. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπερδιπλάσιο πληθυσμό, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα ήταν ένα βάρο που θα μπορούσαμε πιθανότατα να σου σηκώσουμε, άλλωστε αποδείξαμε πέρυσι, όταν είχαμε καθημερινέ ροές πάνω από 7, 8 και 10.000, ότι τα καταφέρναμε. Το κακό είναι ότι δόθηκε χώρο, Δόθηκε χώρο σε ακραία στοιχεία να τορπιλίζουν την κοινωνική συνοχή, να βάλουν κατά τη κοινωνική συνοχή. Και δυστυχώς σε αυτά τα στοιχεία τα ακραία συνεπικουρούν και άνθρωποι, οι πολιτικοί, οι παράγοντες οι οποίοι ανήκουν στο λεγόμενο δημοκρατικό χώρο. Αυτοί οι παράγοντες κινούμενοι από ιδιοτέλεια δεν, ε, νομίζω δεν διστάζουν ε, σε τίποτα, θέλουν να ξεσηκώσουν τον κόσμο και δουλεύουν να ξεσηκώσουν τον κόσμο εξ, στην ουσία αξιοποιώντας ή εκμεταλλευόμενοι το φανατισμό των ακραίων στοιχείων και πολύ φοβάμαι ότι σε ένα σημείο, και το είχα πει δημόσια, ότι αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν να χυθεί αίμα ώστε να δικαιωθούν και να αποκομίσουν τα ωφέλη τα οποία επιδιώκουν. Σήμερα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί, ευτυχώς, και πάλι παρενέβημα και νομίζω ότι κάνανε ένα σημαντικό λάθος. Το λάθος τους ήταν ότι προσπάθησαν να κλείσουν σχολεία και να μην δειχθούν μικρούς πρόσφυγες στο να πάνε να εκπαιδευτούν. Αυτό ήταν το λάθος τους που στην ουσία ξανα, ξύπνησε το ένστικτο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς της τοπικής κοινωνίας και έτσι σήμερα είναι απομονωμένοι. Ελπίζω έτσι να παραμείνουν. Παρακαλώ, έχετε κάποιες ερωτήσεις. Από πλευράς υποσχέσεων που είχαν δοθεί ε, στην ε, ελληνική πλευρά και ενδεχομένως και στο νησί σα ειδικότερα για παροχή βοήθεια και σε προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Frontex κλπ. αλλά και σε τεχνική, υλικοτεχνική υποδομή. Τι έχει γίνει, έχετε κάποια ιδέα, υπάρχουν ελλείψεις, καθυστερήσεις. Θα σας απαντούσα ότι από πέρυσι, από την πρώτη στιγμή όταν αντιμετωπίσαμε την κρίση, ε, εγώ βρισκόμενος απέναντι στην ιστορία λέγοντας ότι είναι το σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας προς εμάς, αυτό που έκανα ήταν ε, να πω ότι θα λειτουργήσω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έξω από τις διαδικασίες δεν αναγκαστήκαμε να κινηθούμε με έναν τρόπο αντισυμβατικό, αλλά ήταν οι καταστάσεις τέτοιες που μας υποχρέωσαν να βδούμε το πρόβλημα και τη λύση και όχι αυτά που μας εμπόδιζαν για να παρέμβουμε. Αυτό έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση. Ε, πήρα πολλές υποσχέσεις, αλήθεια, από την Ευρώπη. Υποσχέσεις που έλεγαν ότι θα ενεργήσει πολύ πιο άμεσα, ότι θα είναι ε, η στήριξη στους Δήμους γιατί και ο Δήμος στην ουσία ανέλαβε είχε αναλάβει όλο το βάρος αλλά στηρίξεις δυστυχώς δεν ήρθαν. Στηρίξεις ήρθαν μόνο από πλευράς της κυβέρνησης με την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Υπουργό αλλά και τους προηγούμενους Υπουργούς και τους άλλους Υπουργούς αλλά όμως η Ελλάδα από μόνη της δεν μπορεί η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να σηκώσει όλο το βάρος για λογαριασμό ολόκληρη της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Θέλει στηρίξει. Άλλωστε η Ελλάδα είναι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι πέραν του ανθρωπιστικού βάρους και τι όποιες προσπάθειες χρειάζεται, χρειάζονται και πόροι. Αυτοί οι πόροι ε, και τι έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν φτάσει ή έφτασαν το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι σήμερα η κατάσταση εξορθολογίζεται και από πλευράς οικονομικής οπότε θα είναι πιο εύκολη η συνέχεια. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Παπαδημούλης, γιατί αποτελεί ένα παραλογισμό. Παραλογισμός είναι όταν ξέρουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι που τις εκφράζουν είναι αυτοί που σηκώνουν το βάρος, είναι αδιανόητο αυτούς να μην τους στηρίζεις, να μην τους χρηματοδοτήσεις ώστε να διευκολυνθούν στη διαχείριση των χώρων που ήδη έχουν, αλλά και στη φιλοξενία των προσώπων που τους ή φιλοξενούμε στα νησιά μας και στις πόλεις μας και αυτά να δίνει στους πόρους σε οργανώσεις ή μη κυβερνητικού ή μεγάλους οργανισμούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας παραλογισμός. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται σε συνθήκες που έχουν υπογραφεί, σε συμφωνίες, αλλά οι συμφωνίες όταν διαπιστώνεις ότι εμπεριέχουν λάθη ε, μπορεί να βελτιώνονται. Υπάρχει λοιπόν ένας σημαντικός λόγος που πρέπει σε αυτό το σημείο να βελτιωθούν οι συμφωνίες όπως και στο άλλο το οποίο επίσης αποτελεί ένα παραλογισμό και φορτώνει τις κοινωνίες των νησιών κυρίως με πρόσθετο βάρος είναι αυτό που λέγεται ότι απαγορεύει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να μετακινηθούν πέραν των νησιών σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας άνθρωποι και να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας στους χώρους αυτούς, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της ίδιας της συμφωνίας. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένας παραλογισμός που πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Άλλωστε η πρόταση που έχω καταθέσει ε, απευθύνεται και στοχεύει, στοχεύει ακριβώς αυτό, τη διάχυση του βάρους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια στην πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, θα ήθελα, Μάρια Ρόνε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημούλη, ε, εν ώψη και συνόδου κορυφ, της συνόδου κορυφής που θα γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή και το μεταναστευτικό είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσουν τις, ε, τα συμφωνηθέντα σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Όπως είπατε και εσείς όμως οι ελλείψεις είναι πολλές και σε τι οφείλεται αυτό, δηλαδή είπατε ότι 10.000 ε, πρόσφυγες είναι έτοιμοι προς μετεγκατάσταση και περιμένουν ε, στην Ελλάδα, αλλά καθυστερεί πολύ αυτό το πρόγραμμα. Ε, επίσης, η Ελλάδα περιμένει στήριξη και σε οικονομικούς πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε τι πιστεύετε ότι οφείλονται όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο ότι κάποιες χώρες ναι, δεν, δεν δέχονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, μήπως είναι και θέμα διαχείρισης. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, Δήμαρχο ε, Λέσβου, ε, μπορείτε να μας πείτε πόσα παιδιά φιλοξενεί, προσφύγων φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Λέσβος ε, και πόσα από αυτά πηγαίνουν στο σχολείο και αν θα θέλατε επίσης να μας πείτε για τους ασυνόδευτους ανήλικες. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ζητάμε και ως ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ως ευρωομάδα της αριστεράς από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν είναι να τιμήσουν την υπογραφή τους, να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Υπάρχει τρομακτική καθυστέρηση και στην υλοποίηση της συμφωνημένου προγράμματος μετεγκατάστασης και στην αποστολή των ειδικών στην Ελλάδα για να υποβοηθήσουν τις διαδικασίες καταγραφής και εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και από πλευράς κρατών μελών. Προφανώς αυτές οι καθυστερήσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούν, κυρία Αρώνη, να αποδοθούν απλώς σε προβλήματα της διοίκησης και της γραφειοκρατίας δείχνουν ένα έλλειμμα πολιτικής βούλησης της ευρωπαϊκής ηγεσία να εφαρμόσει τις αποφάσεις που ήδη έχει πάρει. Το έλλειμμα αυτό είναι τόσο μεγάλο που απειλεί την ίδια την ευρωπαϊκή ενοποίηση με τον κίνδυνο της διάλυσης. Και αυτό δεν είναι μια δήλωση δική μου, είναι μια δήλωση που έκανε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο ίδιος ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Είπε μια Ευρώπη που δεν μπορεί να υλοποιήσει τις αποφάσεις στο προσφυγικό κινδυνεύει με διάλυση. Εγώ αυτό που προσθέτω είναι ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να δουλεύει à la carte. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Όρμπαν ή η κυβέρνηση που στηρίζει ο κύριος Κατσίνσκι στην Πολωνία ή άλλες κυβερνήσεις να θέλουν την Ευρώπη για να παίρνουν κονδύλια για τους αγρότες τους, για τις υποδομές τους, αλλά να αρνούνται να δεχθούν έστω και ένα πρόσφυγα, να στείλουν μια σκηνή, να στείλουν μια κουβέρτα, να στείλουν έναν ειδικό να βοηθήσει η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε όλα τα φόρα και σε όλα τα επίπεδα, όλο ένα και πιο πιεστικά, θα το θέσει και στη Σύνοδο και φυσικά αυτή τη φορά έχοντας πολύ περισσότερα στηρίγματα και συμμαχίες από οποιαδήποτε άλλη φορά. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας από τους συμμάχους της ε, ε, ελληνικής προσπάθειας γιατί με μια πλειοψηφία πάνω από 70% εψήφισε και απαιτεί το αυτονόητο. Να εφαρμοστούν οι αποφάσει για την μετεγκατάσταση. Το ζητούμενο όμω είναι τα λόγια να γίνουν πράξη και σε αυτό ζητάμε τη συνδρομή και των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωση και τη κοινωνία των πολιτών και τη αυτοδιοίκηση και η σημερινή πρωτοβουλία νομίζω ότι σε αυτό στοχεύει να αναδείξει καλέ πρακτικέ και να κινητοποιήσει και τις δυνάμεις της κοινωνίας που είναι κάτω από τις κυβερνήσεις και μπορούν να κάνουν πράγματα για να πιέσουν και τις κυβερνήσεις τους αλλά να βοηθήσουν και τους πρόσφυγες. Κύριε Δήμαρχε. Ε, ακριβή αριθμό κυρία Αρώνη δεν μπορώ να σας δώσω. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητος είναι ότι κανένα παιδί πρόσφυγα, κανένα προσφυγόπουλο δεν θα είναι που είναι στο νησί, δεν θα εμποδιστεί για να πάει στο σχολείο. Όλα τα παιδιά θα πάνε στα σχολεία θα φοιτήσουν και θα φοιτήσουν και θα πάρουν την εκπαίδευση με τον καλύτερο τρόπο. Ε, επίσης να σας πω για τα συνόδευτα ότι πέραν των δομών που σας ανέφερα, τις τρεις δομές, υπάρχουν και άλλες δομές στο νησί, υπάρχουν αρκετές δομές ακόμη, οι οποίες έχουν ανοιχθεί από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες φιλοξενούν ασυνόδευτους ανηλίκους. Θα με επιτρέψετε να, να επισημάνω μόνο προς το πρώτο θέμα της εκπαίδευσης, διότι ακριβώς πήγαν κάποιοι ακραίοι να παρουσιάσουν πρόβλημα στο νησί, κλειδώνοντας κάποιο σχολείο. Και αυτό που τους είπα και τους επεσήμανα και μάλιστα με απόλυτο τρόπο και κατηγορηματικό είναι ότι ασφαλώς το που σας είπα πριν ότι δεν θα μείνει κανένα προσφυγόπουλο το σχολείου αλλά υπενθύμησα ότι μια ακόμα μεγαλύτερη Ελλάδα από αυτή των 10 εκατομμυρίων που ζει στον ελληνικό χώρο ζει στο εξωτερικό. Και αυτή τη Ελλάδος τα παιδιά προοδεύουν, φοιτούν σε σχολεία πηγαίνουν σε πανεπιστήμια και τους δίδονται όλες οι δυνατότητες να προοδεύσουν. Είναι αδιανόητο λοιπόν σε Έλληνα ή σε Ελληναρά να διαμαρτύρεται και να εμποδίζει προσφυγόπουλο να πάει σε σχολείο. Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση, συνάδελφοι. Ναι. Sorry, I'm from the Parliament magazine. Can I just ask what... Κοιτάξτε, ένα-δύο πράγματα να ρωτήσω. Ποια είναι η άποψή σας. Δεν σχετίζεται άμεσα αλλά πώς αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί την κατάσταση στο Καλέ. Οι Βρετανοί δέχτηκαν νέους. Φαίνεται να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τις ηλικίε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Άλλη ερώτηση. Ποια είναι η αποψή σας για τον Βίκτον Ορμπάν στην Ουγγαρία πώς αντιμετωπίζει εκεί το θέμα των προσφύγων υπό το φως του πρόσφατου δημοψηφίσματος. Well, Σας δώσω μια απάντηση. Η θέση της Βρετανίας όσον αφορά τους πρόσφυγες είναι εξωφρενική, εξοργιστική. Αυτοί οι άνθρωποι ξεφεύγουν από το Ισλαμικό κράτος στη Συρία και στο Ιράκ και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Ξέρετε ποιος δημιούργησε αυτό το τέρας, το Ισλαμικό κράτος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βρετανία. Όταν εισέβαλαν το 2003 στο Ιράκ. Και τώρα λένε όχι, όχι. Δεν θέλουμε πρόσφυγες. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε αυτό, καμία σχέση με αυτό. Δεν επομίζονται τις ευθύνες τους. Απλώς λένε ότι οι Έλληνες πρέπει να το φροντίσουν, να κλείνουν τα σύνορα. Είναι μια συμπεριφορά που είναι κατά των νόμων της ανθρωπιάς, της ανθρωπότητας και το σεβασμό ε, της κάθε χώρας και να σέβεται μια χώρα τον εαυτό της. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για όλα αυτά. Αν όχι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και Μεγάλη Βρετανία. Στη ΣΥΠΑ ο Τραμπ λέει, υπόσχεται ότι θα κλείσει όλα τα σύνορα και έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία που ήδη κλείνει τα σύνορα. Μη δεχόμενοι πρόσφυγες. Και τα βασικά επιχειρήματα για το Brexit ήταν ε, οι πρόσφυγες. Το σκέλος της ερώτησής σας που αφορά στην κυβέρνηση Όρμπαν. Η στάση της Ουγγρικής κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Τσαλαπατάει και κουρελιάζει και πετάει στα σκουπίδια όχι μόνο τη συνθήκη της Γενέβης και όσα απορρέουν από αυτή για την προστασία των ετούντων άσυλο, αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Συνόδων Κορυφής για το Προσφυγικό που ο ίδιος ο κύριος Όρμπαν έχει υπογράψει. Είναι μια μεγάλη επιστροφή προς τα πίσω, σε ένα εφιαλτικό παρελθόν όπου η Ήπειρος της Ευρώπης κυριαρχήθηκε από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Και είναι κρίμα γιατί ο ίδιος ο, κύριο, κύριος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι πριν μερικές δεκαετίες εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν σε πολλά άλλα κράτη της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν που λέει ότι όσα κράτη-μέλη αρνούνται να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους για την φιλοξενία προσφύγων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου, οφείλουν τουλάχιστον να πληρώνουν το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο προκειμένου άλλα κράτη να υποδέχονται αυτούς τους πρόσφυγες και να τους φιλοξενούν. Δυστυχώς αυτή η πρόταση της Κομισιόν έχει σκαλώσει στο Συμβούλιο και δεν υλοποιείται, δεν συζητείται για την εφαρμογή της στα σοβαρά. Γι' αυτό λέω πάκτα σουν σερβάντα. Οι συνθήκες, οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Και καλό και τις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να πάψουν να μεταχειρίζονται ευνοϊκά τον κύριο Όρμπαν. Η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δέχεται πιέσεις. Ο κύριος Όρμπαν κάνει τα ίδια ενδεχομένω και χειρότερα, αλλά επειδή ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αντιμετωπίζεται με μια περίεργη ανοχή που φτάνει έως και τα χάδια. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η Ευρώπη, αλλά καρτ. Δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία να ακούνε διαρκώς οι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Και ο κύριος Όρμπαν να τσαλακώνει και να πετάει στα σκουπίδια τους κανόνες και τις κοινέ αποφάσεις. Ε, Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ε, θέλω να σας πω μόνο ότι στη σημερινή διάσκεψη που είχαμε που είχε τίτλο Solid Cities, αλληλέγγυες πόλεις δηλαδή, ο κύριος Γαλινός, ο δήμαρχος ε, της Λέσβου, κατέθεσε μία πρόταση ε, που είναι αυτή, η European Network of Cities, the answer to the refugee crisis το, το δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων, η απάντηση στην κρίση των προσφύγων υπάρχει και στα ελληνικά, υπάρχει και στα ε, αγγλικά ε, και μπορείτε να την, ε, να την προμηθευτείτε και επίσης να παρακολουθήσετε την συνδιάσκεψη που συνεχίζεται στις 2.30 το μεσημέρι ώρα Βρυξελών όπως επίσης ότι όπως και αυτή η συνέντευξη έτσι και η συνδιάσκεψη μεταδίδεται και από το διαδίκτυο ζωντανά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και πολύ και τους διερμηνείς ε, για την ε, βοήθεια πολύτιμη.